Καλημέρα σας. Σας έτοιμοι για την ψηφορία, λέει ο κύριος Ντεκάστρο. Πολύ ωραία. Όπως γνωρίζετε, αναβλήθηκε μία ψηφοφορία, οπότε θα ψηφίσουμε δύο θέματα. Η κυρία Ζωάνα αναβλήθηκε, οπότε η Ριμπέιρο θα είναι η πρώτη ψηφοφορία, το θέμα της κυρίας Ριμπέιρο, και η δεύτερη θα είναι της κυρίας Ανζελίκ Ντελαέ. Εδώ είναι και οι δύο, τις βλέπω. Αν είστε έτοιμοι συναδελφοί τώρα, ε, ε, αν έχετε βάλει τις κάρτες στη θέση τους, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και ξεκινούμε με την συμβαστική υπαριθμόν 1. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Bene, approvato. Andiamo al εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στη συμβαστική 2. Ψηφίζουμε την συμβαστική 2. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε την συμβαστική 3. Ψήφισαν όλοι. Καλώς, συγχαρητήρια. 30 στους 30. Πάμε τώρα στην συμβαστική παριθμών 4. Ψηφίζουμε. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε τώρα. Άρχισε η ψηφορία. Πέρας. Καλώς. Και πάμε τώρα στο 5. Συμβαστική 5. Ψήφισαν όλοι πέρας. Συμβαστική 6. Συμβαστική 6. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 7. Συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. Votato tutti. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 8. Συμβαστική Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 16 του Καπούτο και άλλων. Ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στο 18. Υπέρ. Το 18. Σκοτ. Γκάτο και άλλοι. C'era una richiesta di voto sulla seconda parte, quindi dobbiamo votare. Ζητείτε επιχωριστή ψηφορία για το δεύτερο τμήμα. Για το 18, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να γίνει επαλήθευση ηλεκτρονική. Για το 18.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 υπέρ κατά απορρίπτεται επαλήθευση ηλεκτρονική για το 28 ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 30 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Χάουτουμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε για το 35. Πέρα της ψηφορίας. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με την ίδια διαφορά. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για το 37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά αποχές Καλά, 47 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτωται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το 70 ψηφίζουμε πέρας φορείας. Απορρίπτεται. 71. Όχι, δεν πρέπει να ψηφιστεί. Και πάμε στο 72. Και αυτή του Νέκοφ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά αν συμφωνείτε, επαλήθευση για το 76. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και πάμε τώρα. 79 του Καπούτο, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα θα ψηφίσουμε η τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην συγκέντρια και πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Είναι το θέμα της Ανζελίκ Τελαέ. Ανζελίκ θέλεις το λόγο, όχι. Πάμε να ψηφίσουμε, ωραία. Α, μισό λεπτό. Υπάρχει μια αλλαγή στο συνεργάτες της γραμματείας. Βοτιάμο. Η ετήσια έκθεση που αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Έτοιμοι. Ξεκινούμε από τη συμβαστική 5. Σωστό. Συμβαστική 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Με ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική 4. Ψηφίζουμε το 4. Πέρασε ο Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στη συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Τη συμβαστική 6. Πέρα ψηφοφορία. Και εγκρίνεται συμβαστική. Και τα Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 47. Βιέγκας. Ονομαστική ψηφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Συμβαστική 8. Ηλεκτρονική ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, όχι, συγγνώμη, ο απορρίπτεται. 65. Νταντέν, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68. Μπούντα, υπέρ, σηκώστε το χέρι ευκρινώς υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά κάνουμε επαλήθευση για το 68 ψηφίζουμε πέρας Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 69 ανατασυχηρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται και τώρα συμβιβαστική 9 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 10. Συμβιβαστική 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Νέκοφ. Ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 85 ανάταση χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 97 υπέρ. Σηκώστε το χέρι σας ευγενώς. Νομίζω ότι απορρίπτεται και πάμε στο 98. Ανατασχυρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική παράγραφος και είναι η πρώτη συμβαστική ε, τροπολογία. Συγγνώμη, ψηφίζουμε πρώτη συμβαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επτά, δεν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 ανατάσσει χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εννέα, σκοτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική δύο. ψηφίζουμε Chiusa la votazione. Approvato και εγκρίνεται τροπολογία 11 ανάταση χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 της ισχύτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 20. Ανατασχυρό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφόρια για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Συγχαρητήρια η συγκεντρία. Αντζελή, θέλεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη σύνταξη των συμβαστικών ε, τροπολογιών και χαίρομαι για τους γεωργούς γιατί θα προκύψουν νέες προοπτικές ε, στα θέματα του δικαίου ανταγωνισμού χάρη και σε, αυτό το, σε αυτή την έκθεση και στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε, συγχαρητήρια Αντζέλικ. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σημείο Κοινία, ακρόαση των Επιτροπών Άγκρη και Κοντ είναι δημοσία. Ακρόαση όσον αφορά την ε, εμπειρία από το Λίντερ. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί ε, πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο, ε, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού Προεδρισμού, κυρία Γκρέσλα Γιατί παρακάναμε γρήγορα την ψηφορία, γιατί ακόμα δεν έφτασε η πρόεδρος.